Θα ξεκινήσουμε την απογευματινή μας σύνοδο με την δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της, Ευρω... Ευρωπαϊκής για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σε ό,τι αφορά τη παγκόσμια